Καλό απόγευμα για όλους ε, τους συναδέλφους. Καλώς ήρθατε στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Επιτροπής Προϋπολογισμών πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Είμαι ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και ουσιαστικά είμαι προεδρεύων της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, διότι ο κ. Θεμαγίστρης είναι πλέον δήμαρχος της Νεάπολης στην Ιταλία και δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω τις, ε, τη συγγνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμών που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα το απόγευμα Έχουμε, όπω ξέρετε, στην αρχή μια κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών. Η αρχική ιδέα είναι να είναι εδώ παρόντε και οι δύο πρόεδροι, αλλά δυστυχώ θα προεδρεύω μόνο μου εξ ονόματο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Επομένω, μέχρι τι 4 είναι η κοινή συνεδρίαση Επιτροπή Προπολογισμών και Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Έχουμε δύο ο, την κυρία Γκρέσφετ, τον κύριο Γκερίνη και το πρώτο θέμα που έχουμε ενώπιόν μας είναι φυσικά η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Στο έγκριτο δελτίο κοκομπού Info θα βρείτε τον κατάλογο των γλωσσών για τις οποίες υπάρχει διερμηνία. και ελπίζω ότι έχετε όλη την ε, κάρτα σα, την κάρτα ψηφοφορία, όχι την πιστοτική σα για να ψηφίσουμε. Γιατί θα ψηφίσουμε σε λίγο και η ψηφοφορία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική. Αυτή η συνεδρία μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Ζωντανή. Εάν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο το οποίο βρίσκεται αριστερά σα, θα είσαστε γκρο πλάν στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Θέλω να μεταφέρω επίση και τη συγγνώμη πολλών συναδέλφων μα, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι παρόντε επειδή ένα από τα πρώτα θέματα είναι η έγκριση προηγουμένων, πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, θα ακολουθήσουμε τη συνηθισμένη διαδικασία μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση. Αν έχετε κάποιε ενστάσει, να τι καταθέσετε. Παρακαλώ. Θέλει κάποιο να κάνει κάποια σχόλια. Παρακαλώ. Σε προσωπικό επίπεδο, λέει ο κύριο Σοντή, αυτή τη βδομάδα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τη ζώνη του ευρώ υπέγραψαν μια συνθήκη για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Έχω λάβει γνώση αυτού του εγγράφου. Εδώ δεν υπάρχει καμία απολύτως διάταξη δημοσιονομικού ελέγχου, καμία διάταξη κοινοβουλευτικού και πολιτικού ελέγχου. Υπάρχουν μονάχα η δυνατότητα παρέμβασης ιδιωτικών εταιριών λογιστικού ελέγχου. Εκτιμώ την ικανότητα των εξωτερικών ελεγκτών αλλά ξέρω ότι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ένα εθνικό ελεκτικό συνέδριο ή ένα ευρωπαϊκό ελεκτικό συνέδριο ή ένα κοινοβούλιο δεν εμπλέκονται. Ο ρόλος των κοινοβουλίων είναι να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Έχουμε ένα μηχανισμό με 700 ή 800 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα στο οποίο μηχανισμό δεν υπάρχει έλεγχο ούτε από ελεγκτικό συνέδριο, ούτε από Εθνικό Κοινοβούλιο, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα άπρεπη αυτή η απόφαση η οποία έχει ληφθεί. Ευχαριστώ κύριε Όντι. Είδατε ότι υπήρξε υποστήριξη από τους συνοδεύτρες. Κύριε Ρίμπερ και εσείς για το ίδιο θέμα ή κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να παρατηρήσω ότι το Κοινοβούλιο έχει κάποιους κανονισμούς καινούριου τώρα στο επίπεδο του lobbying, την ε, παρουσία των ομάδων πιέσεων αυτό το βρίσκω πολύ θετικό και είχαμε κάνει και μια ακρόαση εδώ για το λεγόμενο whistleblowing, τις καταγγελίες και από αυτή την ακρόαση ήλθε μια νέα ιδέα να έχουμε ένα ενίο καθεστώ για τι Ευρωπαϊκέ Ενώσει. Θα ήταν χρήσιμο η δική μα Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλία για ένα ενίο καθεστώ των Ευρωπαϊκών Ενώσεων, γιατί πιστεύω στον τομέα αυτό να εξασφαλίσουμε κάποιε προδιαγραφέ ε, ε, διαφάνειες και να τα θέσουμε όλα αυτά σε μια σαφή νομική βάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να το αντιμετωπίσουμε αυτό στη συνεδρία των συντονιστών. Ο κύριος Μίλτερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Οντί το θέμα όμως το οποίο πρέπει να θέσουμε είναι τι ελπίζουμε να πετύχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά τα θέματα. Μία επιλογή θα ήταν να ζητήσουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ίσως στην επόμενη συνεδριασή μας μπορούμε να συζητήσουμε αυτή τη νομική γνωμοδότηση, τη νομική γνωμοδότηση για να μπορέσουμε να διακριβώσουμε τι ακριβώς εξουσίες έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ Γιάννη για την τόσο επικοδομητική αυτή πρόταση. Ο κ. Ριβελίνη. Όχι, Πρόεδρε. Για άλλο σημείο παίρνω το λόγο. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή. Και αυτές τις εβδομάδες και τους μήνες δουλεύει επί κάποιων θεμάτων και φακέλων που είναι πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι περίεργο που ο κύριος Δεμαγκίστρης που εδώ και πάνω από δύο μήνες έχει εκλεγεί δήμαρχος δεν έχει ακόμα υποβάλει την παρέτησή του από, Ευρω... από Ευρωβουλευτής. Από ό,τι ξέρω, τέλος Ιουνίου έπαιξε το ρόλο της Επιτροπής Κοκομπού. Ε, εμφανίστηκε δηλαδή με αυτή την επίσημη ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ζητήστε από τον συνάδελφο ή πρώην συνάδελφο τέλος πάντων να αποφασίσει τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Δεν μπορεί να έχει ε, δύο ιδιότητες. Δεν γίνεται. Ε, ο, εσείς λοιπόν ως πρόεδρος α, θα πρέπει να του πείτε ότι εκείνος δεν μπορεί να συγχύσει να κατέχει μια θέση η οποία στην πραγματικότητα χειρεύει. Ε, er ε, Ευχαριστώ. Ε, σημειώνουμε την παρατήρησή σας. Εμείς ε, στην ομάδα μας, στην ομάδα των φιλελεύθερων, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Θα ξεκαθαρίσουμε, ελπίζω, τα πράγματα στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού το Σεπτέμβριο. Ούτω ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με φυσιολογικό τρόπο τις συνεδριάσεις Για τα πρακτικά, ο κύριος ε, Μούλντερ ζήτησε να προσφύγουμε στην νομική υπηρεσία για να μας δώσει μια γνωμοδότηση. Αν συμφωνούν οι συνάδελφοι λοιπόν επίσημα, θα ήθελα να αποφασίσουμε να προσφύγουμε όντω στην ε, νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για να δούμε τι άποψη έχει. Συμφωνούμε, η κυρία Γκρέσλερ. Ακριβώ. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό και είναι εγγύηση των πρώτων 60 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προπολογισμό του. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίσω σε ποιο βαθμό εμεί μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά τα ποσά στο επίπεδο των 61 δισεκατομμυρίων και πώ μπορούμε να ε, κινητοποιηθούμε. σω ο Γενικό Διευθυντή από την Υπηρεσία των Προπολογισμών μπορεί να μα δώσει κάποιε διευκρινήσει. Ευχαριστώ. Er Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα λοιπόν εδώ προς την Επιτροπή. Μπορώ να σας δώσω το λόγο, Επιτροπή, για να απαντήσει την κυρία Γκρέσλερ, ο κύριο Ταβέρνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου. Αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Τα 60 δισεκατομμύρια για τα οποία έκανε λόγο η κυρία Γκρέσλερ ε, για αυτά. Ε, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στο σημείωμα ε, για τα λογιστικά. Δεν το έχετε, αλλά θα φτάσουν. θα το υπογράψω αύριο ή μεθαύριο. Και όλες οι πληροφορίες και όλες οι κινήσεις μέχρι τη στιγμή που υπογράφω υπάρχουν σε, αυτή την, σε αυτό το σημείωμα για τους λογαριασμούς. Ε, λίγες μέρες υπομονή και θα έχετε όλες αυτές τις α, πληροφορίες. Αλλά αυτά ε, είναι άλλη ιστορία από αυτά που λέει ο κ. Σοντή. Ο κύριος Σοντή μιλάει για τον, το διακυβερνητικό θέμα. Έτσι. Ε, απαντάω λοιπόν στην κυρία Γκρέσλερ. Ε, δεν απαντάω στον κύριο Ντί. Επιφυλάσσουμε για αυτό το θέμα. Ναι. Ημέν, το πρώτο, οι δεν το επιτρέπουν. Γι αυτό, δεν το παραλείπουν. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να συζητήσουμε πολύ πιο σοβαρά τι θα κάνουμε με αυτά τα 60 δις ευρώ, σε ποιο βαθμό δηλαδή αυτά τα ποσά ε, είναι ε, ποσά που διατίθεται με υποχρέωση λογοδοσίας και ποια είναι η κατάσταση μέχρι τώρα στη διάθεση των ποσών αυτών μέχρι σήμερα 13 Ιουλίου 2011. Δεν έχουν κινητοποιηθεί παρά μόνο μέσω μέτρων back to back όπως τα λέμε. Δηλαδή αυτό που κάναμε είναι κάποια δάνεια με ίδιους όρους εκτός για την Ιρλανδία, όπου υπήρχε ένα περιθώριο ε, στις αρχές του 2011. Ο προϋπολογισμός ούτως ή άλλως κινητοποιείται μόνο σε περίπτωση χρεοκοπίας. Οι αρχικές λοιπόν στις αρχικές φάσεις δεν κινητοποιούμε, δεν προσφεύγουμε στον προπολογισμό. Ούτως Ούτε η όλες αυτη πολύ γρήγορα ε, περιπλέκεται. Και καλό είναι να έχετε κείμενα για να έχετε κάποιες πληροφορίες, ώστε να μιλήσετε με τα λόγου γνώσεως και να θέσετε και λεπτομερείς ερωτήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μάλιστα συντομότατα. Eh, μάλιστα. Σημειώνω την πρόταση του κ. Ταβέρν, δηλαδή να μας υποβάλει αυτό το έγγραφο και αρχές Σεπτεμβρίου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να με το σημείο αυτό τον 60 δις. Έγινε σχεδόν σημείο από τα διάφορα αυτό το σημείο. Έχετε και άλλες παρατηρήσεις τέλος πάντων. Όχι. Πάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Δημοσιονομικός κανονισμός. Με τους δύο εισηγητές τον κύριο Ριβελίνη και την κυρία Γκρέσλερ. Είχαμε προβλέψει αρχικά να δούμε τις τροπολογίες. Πολλές ομάδες, λόγω της περιπλοκότητας της ψηφοφορίας και λόγω του ότι κάποια πράγματα ε, είναι ασαφή, να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Κάποια στιγμή θα ψηφίσουμε, λοιπόν, το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω πότε ακριβώ. Προς το πρώτο δεν έχουμε βρει ημερομηνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπου και οι δύο εισηγητέ θα μπορούσαν να βρεθούν ταυτόχρονα στι συνεδρίε. Ψάχνουν αυτή τη μαγική ημερομηνία. Τέλο πάντων, το Σεπτέμβριο πάντω θα ψηφίσουμε αυτό το θέμα. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή συζήτηση. Σα προτείνω να δώσουμε το λόγο στου δύο συνεισηγητέ αν το επιθυμούν. Αν όχι, οι συνάδελφοι μπορούν να θέσουν ερωτήσει. Ο κ. Ζιβελίνη θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εφόσον μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο, θα ήθελα να, κάνω, να παρουσιάσω ένα προβληματισμό για τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπει ο κανονισμός. Αυτά τα μέσα είναι το πιο σημαντικό θέμα, το πιο ενδιαφέρον θέμα για, του κανονισμού. Λόγω και όλων όσων συμβαίνουν αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες στην παλιά μας, στη γυραιά Ευρώπη. Η πρόταση της Κομισιόν ε, αφορά κυρίως δύο άρθρα, το 130 και 131 του Δημοσιονομικού ε, Κανονισμού και το 39 C ε, έως το 39 D ε, των εφαρμοστικών διατάξεων. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα μέσα. Ποια είναι τέλος πάντων αυτά τα μέσα. Το άρθρο 130 τελικά ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Πρόκειται για μέτρα ε, χρηματοδοτικής υποστήριξης της Ένωσης που βαραίνουν το προπολογισμό με στόχο να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι, αλλά συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι, χάρη σε κάποια μέσα όπω τα δάνεια, οι εγγυήσει, ε, επενδύσεις ή ε, συμμετοχές μετοχικού χαρακτήρα ή ιονή μετοχικού χαρακτήρα ή μέσα, μέτρα μάλλον, που ε, συνδέονται με επιδοτήσεις. Αυτά τα μέσα σε πολλές περιπτώσεις καλύπτονται, αφορούν πολιετή προγράμματα και για να συλλέξει κονδύλια η Κομισιόν θα εκδώσει τα λεγόμενα project bonds, τα ομόλογα έργων. Η Κομισιόν προτείνει να ασχοληθεί κυρίως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με αυτό το θέμα, η οποία και με βάση στα 308 και 309 άρθρα της συνθήκης θα έχει μία ειδική αποστολή. Θα είναι το όργανο το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ε, δεν μπορεί να, θα μπορεί να κάνει επίσης ε, διαγωνισμούς και θα μπορεί να υποβάλει προτάσεις για την ε, χορήγηση αυτών των επιδοτήσεων. Οι εισηγητές θεωρούν ότι αυτή η προσέγγιση είναι αποδεκτή, αλλά νομίζω ότι η Κομισιόν έχει το καθήκον να μας ε, παρουσιάσει και άλλες διευκρινήσεις. Πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα μείζον πρόβλημα στην πρόταση της Κομισιόν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να εκχωρήσει την αρμοδιότητα ε, εκτέλεσης σε μία από τις θηγατρικές της, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να εμπλακεί το Κοινοβούλιο η δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων, μην ξεχνάτε ότι είναι εντελώς ανεξάρτητη. Αν όλα αυτά τα δεχτούμε, τότε οι μηχανισμοί ελέγχου δεν θα είναι στα χέρια πια του Κοινοβουλίου. Ξεφεύγουν από τα δικά μας χέρια, αλλά θα βασίζονται σε συμφωνίες που συνάπτει η ίδια ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, άρθρο 308 ΤΕΡ παράγραφος 1 και 2. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτά τα μέτρα και να ζητήσουμε τα εξή. Να εξορθολογήσουμε σε σχέση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην δημιουργούμε αντιφάσεις ανάμεσα ε, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού από τα κράτη-μέλη και στην εκτέλεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο, να εξασφαλίσουμε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κατάλληλο ρόλο στη φάση της εκτέλεσης, ούτως ώστε να μπορεί να επαληθεύει την υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων. Τρίτον, να μην δεχτούμε μια αποκλειστική μεταχείριση που θα αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα κάνει ό,τι θέλει μόνη της, παρά τα όσα λέει η συνθήκη. Τέταρτον, να εξασφαλίσουμε ότι οι μελλοντικές εκχωρήσεις και αναθέσεις θα γίνονται μόνο στο πλαίσιο μια συγκεκριμένης νομικής βάσης. Πέμπτον, να διατηρήσουμε την ευθύνη της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τέλος, αυτές τις μέρες ήρθα σε επαφή με κάποιους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και με άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Και νομίζω ότι ο χρηματοδοτικός ε, κανονισμός και εκεί που μιλάει, μιλάει συγκεκριμένα για τα χρηματοδοτικά μέσα, εκεί θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιες αλλαγές. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορεί να έχει αυτή την προνομιούχα σχέση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μια μεγαλύτερη εμπλοκή των ε, ταμιευτηρίων, που συχνά Ε, προβλέπουν καλύτερους όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε στο εσωτερικό των, δημο... χρηματοδοτικών αυτών μέσων την υποχρέωση να εμπλέκονται και οι περιφέρειες των κρατών μελών. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ξεκινώντας από τα χρηματοδοτικά μέσα αυτού του κανονισμού. Περιμένω ερωτήσεις από τους συναδέλφους και ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ, λέω και ο Πρόεδρος. Κυρία Γκρέσλε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους σοσιαλιστές συναδέλφους να μας δώσουν την άποψή τους για τις κατεχώρηση ή κατεξουσιοδότηση πράξης. Στον κύριο Ρεβε... Ριβελίνη, νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πάλι τα θέματα της ισοδικίας στα χρηματοοικονομικά. Πολλοί συνάδελφοι έχουν απογοητευτεί από το γεγονός αυτό, γιατί είχαμε, εργαστεί τα θέματα, είχαμε επεξεργαστεί τα θέματα αυτά πάρα πολύ και υπήρξε πριν από δύο εβδομάδες μια συν, μια ακρόαση του ΕΛΚ με συναδέλφου από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και τα περιφερειακά θέματα και έμαθα πολλά πράγματα. Υπάρχει το πρόβλημα στα εργαλεία αυτά τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό υποαπορροφούνται. Ο καθένα έχει δημιουργήσει το δικό του επί τούτου μοντέλο. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τον έλεγχο τον οικονομικό και θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ένα κοινό επίπεδο για όλα αυτά. και σε χώρες όπως η Τσεχία έχουμε μία μόχλευση 2,2 έως 3 ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πολύ λίγο. Συγγνώμη, στα προγράμματα Τζέρεμι και Τζέσικα, συγγνώμη, στην Τσεχία έχουμε μόχλευση 2,2 έως 3. Και μπορώ να πω ότι η Σικελία και η Καμπανία και συγχαίρω τον κύριο Ριβελίνη είναι από τις περιοχές όπου υπήρξε η καλύτερη απορρόφηση. Ξέρουμε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι ακόμα ασαφής. Περιμένουμε την ε, έκθεση της Κομισιόν, δεν ξέρουμε ακόμα και ποια είναι η θέση της Κομισιόν για όλα αυτά τα ζητήματα. Μετά από αυτήν λοιπόν την, ε, μετά από αυτή τη συζήτηση και με την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου που ήταν πάρα πολύ θετική, νομίζω ότι θέσουμε, πρέπει να θέσουμε και πολλά ακόμα ερωτήματα για το αν φτάνουν πραγματικά στους αποδέκτες τα χρήματα. Και τι γίνεται όταν τα χρήματα αυτά επανέρχονται. Είναι αυτή τη στιγμή όμως μια κατάσταση ότι ο καθένας θεωρεί ότι όλοι παίρνουν χρήματα εκτός από τον ίδιο και δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια. Τι θα γίνει επίσης με ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο προβλέπει επενδύσεις οι οποίες ξεπερνούν τη δημοσιονομική περίοδο και τι θα γίνει και με τον τελικό αποδέκτη. Ο αποδέκτης είναι το ταμείο αυτό, αρκεί να πάρει χρήματα λοιπόν το ταμείο αυτό ή πρέπει τα χρήματα αυτά να μπουν σε κάποιο σχέδιο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα ταμείο ο τελικός αποδέκτης. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να οδηγηθούν σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Αλλιώ θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει με τα χρήματα αυτά και αν πρέπει να επανέλθουν. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και προσεκτικά επομένω. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν να μας δώσει επικαιροποιημένα σημεία και στοιχεία για να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε να έχουμε μια καλύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτά τα οποία μας έχει πει το ελεγκτικό συνέδριο με την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει για το 2010 γιατί τα πράγματα δεν φαίνεται ότι έχουν γίνει με τον καλύτερο τρόπο αλλά σας ε, ζητώ και πάλι και επιμένω να υπάρξει πραγματικά μια επικαιροποίηση για όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το διοικητικό κόστος, πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει, να υπάρχει μια διαδικασία παροχής αναφορών στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τη λεγόμενη μόχλευση σε σχέση με την ε, ε, αποδοτικότητα αυτών των μέτρων και τους ελοχεύοντες κινδύνους. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Βλέπετε τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες από τη σελίδα 46 υπάρχουν νέες προτάσεις για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Για τις πράξεις αυτές έχουμε στον πίνακα αυτά αυτό πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό είναι το έγγραφο εργασίας που αφορά το, τη λεγόμενη κοινή συμφωνία ή κοινή κατανόηση. Μου λέει τώρα η νομική επιτροπή ότι δεν έχει περάσει ποτέ αυτή η κοινή ε, συμφωνία, το, το common understanding, δεν έχει επομένως νομικό χαρακτήρα, δεν έχει περάσει ποτέ από την ε, Ολομέλεια. Πρέπει όμως να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή νομική βάση. Εμείς θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της εκχώρησης και της επανεκχώρησης εξουσιών. Αυτό για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπου υπάρχουν προβλήματα, για να ξέρουμε ότι σε περιπτώσεις όπως αυτές του προϋπολογισμού να υπάρχουν σαφείς εκχωρήσεις εξουσιών. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι ότι υπάρχουν πάντα πράξεις κατεχώρησης όταν πρέπει να αναλάβει κάποιες εξουσίες η Κομισιόν. Εμείς έχουμε αποκλίνει λιγάκι από την αρχική μας διαπραγματευτική θέση. Αν συνεχίσουμε να αποκλίνουμε τόσο πολύ δεν έχει νόημα καν να διαπραγματευόμαστε. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παραμείνει πιστό στο πνεύμα της συνθήκης Λισαβόνας και να κάνει μια διάκριση μεταξύ αυτού που είναι σημαντικό και αυτό που δεν είναι σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε την ήρα από το στάρι και να διατηρήσουμε τις ευθύνες μας και να προτείνουμε και στην Κομισιόν μια διαδικασία για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι κατεχώρηση, οι μάλλον πράξεις, ώστε να μπορούμε να έχουμε σαφείς τέτοιες πράξεις οι οποίες διατηρούν και τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ορισμένε περιπτώσει έχουμε αποκλίνει από αυτέ τι διαδικασίε, αλλά είναι απαραίτητο για λόγου διαπραγματευτική ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντί τη Κομισιόν και του Συμβουλίου να έχει μια σαφή θέση. Για τι μεταφορέ πιστώσεων, θα ήθελα να σα αναφέρω ότι οι τροποποίησει τη Κομισιόν ξεπερνούν αυτά που είχαν συμφωνηθεί το 2009 στη διαδικασία του προπολογισμού. Αυτά ουσιαστικά ακυρώνουν ορισμένα τμήματα του προπολογισμού. Εμείς θελήσαμε να πλησιάσουμε την ε, Κομισιόν και να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία, όπως παραγωγικά σε θέματα τα οποία είχαν γλωσσικό χαρακτήρα, αλλά υπήρχαν σε πολλές περιπτώσεις ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν από ένα τομέα σε ένα άλλο. Γι' αυτό ο στόχος μας ήταν εκεί που υπήρχαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων να τις συγκεράσουμε κατά κάποιο τρόπο εγώ θεωρώ ότι η διαδικασία του προπολογισμού δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα παραλογισμό. Θα πρέπει εμείς να κρατήσουμε τις εξουσίες μας μέσα στη διαδικασία του προπολογισμού και γι' αυτό εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε και ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, ίσως 7 ετών, σε σχέση με το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται ο προϋπολογισμός. Έχουμε προσπαθήσει να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις είναι απαραίτητο όμως να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα οποία είναι εφικτά και όχι σε αυτά τα οποία μπορεί να αλλάξουν. Γι' αυτό τονίζω τη σημασία αυτών των ε, συμβαστικών τροπολογιών θα είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τον κατάλογο ψηφοφοριών. Φυσικά αυτό θα γίνει μετά τι διακοπέ, αλλά θα επανέλθουμε και σε αυτή τη χρονική στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Δύο να πάρουν λόγο. Ο κύριο Φέρμ και κυρία Μπράντνερ. Κύριο Κανένα άλλο. Τρία άτομα τελικά. Ο κύριος Φέρμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους συζητητά για την αφοσίωση με την οποία επιτέλεσαν το έργο τους. Είναι δύσκολο το υλικό που έχω αναλάβει και ξέρω ότι προσπαθούν να εξασφαλίσουν συμβαστικές λύσεις μεταξύ των ομάδων. Αλλά έχω τα εξή ερωτηματικά για τα δημοσιονομικά μέσα καταρχάς κύριος Κάλφιν δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά με παρακάλεσε να κάνω εκ μέρους του συντονιστή της ε, εκτέξης σχόλια. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με εκτέλεση προϋπολογισμού και τις ε, προτάσεις αυτές, ε, θα υπάρχει όντως περιορισμός του της έκτασης του ελέγχου και της δυνατότητας να αξιοποιήσουμε τα ποσά αυτά για την υποστήριξη συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Παρακάλεσε ο συνάδελφος να τα επαναφέρω τα θέματα αυτά γιατί τελικά φοβάται ότι μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία της συμπράξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Επίσης μια ερώτηση για την κυρία Κρέσλε που την έχουμε ξανασυζητήσει εντωμεταξύ. μεταξύ η πρόθεση σας ποια είναι. Ενδεχόμενη αναβολή θα οδηγούσε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο και στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Ε, τι προτίθεστε όμως να κάνετε, θέλετε μια ε, διαδικασία πλήρους πρώτης ανάγνωσης με ψήφισμα, να γίνει δηλαδή ουσιαστικά όλη η συζήτηση και οι δηλώσεις ή θέλετε να το περιορίσετε σε μια συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας και για λόγους διαφάνειας παρακαλώ εγώ προσωπικώς να γίνει η πλήρης διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης για να περάσει το θέμα μετά στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Επίσης με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της ε, διαφάνειας, το οποίο ξέρουμε ότι είναι μάλλον δύσκολο ζήτημα. Προσπαθούμε να διακρίνουμε μεταξύ μεταφορών που μπορεί να έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία και μεταφορών ή ε, εμβασμάτων που μπορεί να έχουν σαν στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής και την ε, πιο ευέλικτη λειτουργία του προπολογισμού, χωρίς όμως σημαντικέ πολιτικές επιπτώσεις. Εδώ και 19 μήνες όμως και από τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη έχουμε διαφορετικούς κανόνες ενισχύει από ό,τι στο παρελθόν και φαίνεται ότι έχουν φέρει ε, καλά αποτελέσματα αυτοί οι κανόνες. Τώρα όμως οι μας παρακαλούν να οπισθοδρομήσουμε δεν δέχονται δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για, τις, για τα εμβάσματα εκείνα που έχουν πολιτικό χαρακτήρα και άλλοι για εκείνα που έχουν μάλλον τεχνικό χαρακτήρα. Και ερωτώ τους φυσικητές εάν θεωρούν όντω ότι είναι ε, φρόνιμη μια τέτοια ε, επιλογή. Με τη δουλειά που έχουμε. Είμαστε διατεθειμένοι για κάθε αίτημα να ζητούμε πιο πολλές πληροφορίες ε, ακόμα και για ποσά τα οποία θα έχουν πολιτική επίπτωση. Αυτό έχει πράγματι πιστεύετε ε, σαν αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση του στόχου της απλούστευσης, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ε, προσπαθήσετε κι εσείς να βοηθήσετε να βρούμε μια συμβαστική λύση για τις μη πολιτικά σημαντικές μεταφορές κονδυλίων. Για τις κατεξουσιοδότηση πράξη επίσης, τα σχόλια των εισηγητών και το επιβεβαιώνει και η κυρία Γκρέσλε προφορικός. Ε, τα γραπτά σχόλια πάντως βλέπω ότι τροποποιούν το χαρακτήρα της ε, συνεννόησης του ε, μνημονίου συνεννόησης με τον περιορισμό παραδείγματι του χρόνου εξέταση για τι αντιπροσωπίε. Και με συγκλονίζει αυτό, διότι αν δεν απατώμε μόνο ένα χρόνο έχει περάσει από εκείνο το μνημόνιο συνεννόηση. και δεν καταλαβαίνω πώ είναι δυνατόν να τροποποιούμε επί τη ουσία αυτέ τι προτάσει χωρί συνένεση των πολιτικών ομάδων και εκείνων οι οποίοι είχαν αναλάβει τη διαπραγμάτευση επί των κατεξουσδότηση πράξεων την εποχή εκείνη. Γιατί αυτό εάν ε, μείνει του, πιστεύω ότι ουσιαστικά ανατρέπει την πολιτική ισορροπία που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και ει ε, προσυμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να απαντήσει, παρακαλώ σε όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Φέρμε, κυρία Μπραντνερ, ως εισηγήτρια για γνωμοδότηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους εισηγητάς και κυρίως την κυρία Γκρέσλε Θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας ε, θεωρεί εύστοχη την νέα διατύπωση του ποσοστού σφάλματος, του κινδύνου σφάλματος. Για το ζήτημα των ε, εμβασμάτων συμφωνούμε με τον κύριο Φέρμα. Για, το, για τους τομείς στους οποίους θα έπρεπε να εμπλεκόμεθα για έλεγχο και σε ποιους όχι. Ε, αν θα πρέπει να επεξεργαστεί ενδεχομένω και νομίζω ότι θα ήταν ε, σκόπιμο ούτως ή άλλως να γίνει συζήτηση στο θέμα αυτό ευρύτερα για να <clears throat> ξαναδούμε όλοι και να υπενθυμίσουμε τις θέσεις μας. Για το θέμα της διαφάνειας ο συμβασμό, από ό,τι βλέπω συνεπάγεται ότι θα επαναπροσδοριστούν πολλά πράγματα σε κάθε τομέα χωριστά. Αυτό σημαίνει ότι στου ορισμένους τομείς ε, δεν θα έχουμε ιδιαίτερη πρόοδος προς τη διαφάνεια, ίσω και μηδενική, ενώ από την άλλη μπορεί να εξασφαλίσουμε κάποια διαφάνεια σε κάποιου τομείς, ενώ παράλληλα την παρετούμαστε από την ιδέα της διαφάνειας σε άλλους, όπως Φερρυπίν της Γεωργίας. Ερωτώ λοιπόν γιατί το προτείνετε αυτό. Θεωρείτε ότι δεν θα μπορέσετε να τηρήσετε τις προδιαγραφές ε, διαφάνειας στον τομέα της Γεωργίας και γι' αυτό προτιμάτε να, τους, να τη διαφυλάξετε, τουλάχιστον να διαφυλάξετε τους όρους της διαφάνειας στους άλλους τομείς ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι. Για δε τον κατάλογο ψηφοριών, στο άρθρο 34 θα ήθελα να κάνω μια διορθώση. Μιλάτε για τροπολογία 48 και ε, λέτε ότι είναι ταυτόσιμη με την τροπολογία της άφετη ε, παριθμών 3. Δεν είναι ταυτόσιμες, είναι πολύ σημαντική. Η διαφορά για μας έχει να κάνει με τα δεδομένα που αφορούν το φύλλο. Δύο λέξεις κάνουν όλη τη διαφορά και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πιστεύω αυτό. Ή δεχθείτε τις δύο αυτές λέξεις ή πάντως μη δεχθείτε ότι είναι ταυτόσιμες ε, οι δύο τροπολογίες. Επίσης, τροπολογία τη δική σας 375 για τις ανθρωπιστικές ε, κρίσεις και τις κατεπίγουσες περιπτώσεις. Υπάρχει μια σχετική τροπολογία υπαριθμών 11 της ΑΦΕΤ, η οποία θα προβλέπετε από τον κατάλογό σας να ψηφιστεί μετά από τη δική σας. Όμως είναι ευρύτερο το πεδίο της και ίσως θα έπρεπε να προηγηθεί της δικής σας τροπολογίας παριθμών 375 ή 11 της ΑΦΕΤ. Αυτό όμως είναι θέμα μάλλον τεχνικό. Και επίσης στο άρθρο 54 η σύγκρουση συμφερόντων δίνεται ως αιτιολόγηση τους εφαρμοστικούς κανόνες όπου επαληθεύσαμε εμείς και διαπιστώσαμε ότι δεν ισχύει αυτό, δηλαδή δεν επαρκούν οι εφαρμοστικοί κανόνες. Ρωτώ λοιπόν τι ε, λόγο σας όθησε σε αυτή την αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάιερ, ο κύριος Γκάιερ έχει το λόγο. Όχι Φραντσίσκα, Φραντσέσκα είναι συνάδελφος. Ρεπιπτόντος. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να ξαναζητήσουμε τα θέματα αυτά. Με μεγάλη χαρά ε, ξανάρχομαι στη συζήτηση αυτή. Δεν έχει συμφωνήσει στην ψηφοφορία η δική μας ομάδα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πιστεύω θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και να διαφωτίσουμε τις συνέπειες που μπορεί να έχουν. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια πρακτική παρατήρηση για τα δημοσιονομικά μέσα. Θα πρέπει νομίζω να αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε εν τέλει να επιτύχουμε. Δύο χρόνια μόνο έχω στο Κοινοβούλιο και δεν είχα καμία πρόθεση να ε, αναλάβω δραστηριότητα ελέγχου του προπολογισμού εξάπαντος ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά είχα από την επαγγελματική μου πρώτερη δράση μεγάλη εμπειρία από τις συμπράξει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και στη Γερμανία υπήρχε ένα ζήτημα μεγάλο ως προς ε, τον έλεγχο αυτού του προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν σε ένα τέτοιο σχέδιο είχε συμφωνηθεί ότι ο ιδιωτικός παράγων ε, συμμετέχει σε τέτοια σύμπραξη μόνο εφόσον είναι υπεύθυνο, ενέχεται δηλαδή σε υποχρέωση, αλλά και αποφέρει κέρδος. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει αυτή η συμμετοχή του ιδιωτικού επενδυτή. Εάν θέλουμε λοιπόν ε, ΣΔΙΠ και θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους ρυθμίσεις το να έχουμε κάνει μια ρύθμιση και να έχουμε μια προπόθεση, μια πρόθεση, θα πρέπει αυτή τουλάχιστον να ρυθμίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδάλω δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί ποτέ και να ισχύσει ΣΔΙΔ, ΣΔΙΠ, γιατί κανένα δότη επενδυτή δεν θα θέλει να συμμετάσχει σε αυτήν. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε ελκυστικές αυτές οι πράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσα από τις δυνατότητες ρύθμισης αυτών των σχεδίων. Και επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτές οι ΣΔΙΤ δεν, είναι, ε, δεν έχουν ταχεία λειτουργία και εξέλιξη. Τουναντίον είναι βραδία εξέλιξη η συμπράξη δημόσιου και τομέα. Γιατί, τουλάχιστον όσον αφορά το γερμανικό δίκαιο, όταν πρέπει να έχουν διαλευκανθεί και ρυθμιστεί όλα τα ζητήματα τη ενοχή, τη ευθύνη, ε, και ούτω καθεξής που προβλέπονται για τον ιδιωτικό επενδυτή εκ των προτέρων μέχρι να προχωρήσει η υλοποίηση αυτή η σύμπραξη έχει περάσει πολύ καιρό. άρα προφανώς θα πρέπει να υπάρχει το θέλγητρο του κέρδους που θα αποκομίσει ο ιδιώτης επενδυτής για να μπορέσει να μείνει μέσα σε μια τέτοια σύμπραξη. Είναι λάθος και ψευδές ιστρονομήσει κανείς ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα μέσα από μια σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα. Μπορεί να προχωρήσει πιο οικονομικά. Μπορεί να κερδίσει δηλαδή σε ε, πόρους και σε οικονομία κλίμακα, αλλά σε τίποτε άλλο, όχι σε χρόνο πάντως. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το ζήτημα βέβαια μετά τη αρμοδιότητας των εντοπίων δικαστηρίων σε κάθε περίπτωση, όταν και αν προκύψει κάποιο ζήτημα, κάποια διαφορά. Αυτό το επισημαίνω διότι υπάρχει διπλός κίνδυνος και να είναι λάθος η επιλογή και να μην λειτουργήσει όπως πρέπει το σχέδιο. Η επιλογή δηλαδή να έχει γίνει εσφαλμένα. Επίσης θέλω να σημειώσω την υποστήριξη μας ως προς τη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 8. Ειλικρινά το λέμε αυτό. Αλλά πηγαίνοντα από τα πίσω προ τα μπρο, Στο σημείο 2, στην παράγραφο 7, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνω. Στο πρώτο ήμιση, στο ζήτημα των ε, ποσών που αναφέρονται. Αυτά δεν είναι τα ποσά που μέχρι τώρα δεν έχουν κρέψει από τον προπολογισμό. Αυτό δεν εννοεί το κείμενο. Αν είναι έτσι να το δεχθώ, γιατί βέβαια θα ήθελα ό,τι λεφτά δεν έχουν απορροφηθεί να επανέρχονται στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Στο δεύτερο ήμιση, Εκεί που, λέει, που ξεκινάει με το in case no budgetary appropriations, εάν δεν μπορούν να εντοπιστούν δημοσιονομικά ποσά, ε, οι πόροι δημοσιονομικοί κτλ. Ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό συνάδει με τη συνθήκη. Γιατί καταλαβαίνω, πολιτική βούληση δεν, ε, δεν λείπει. Στο σημείο 2 της παραγράφου υπαριθμών 7 και βοηθάει και το άλλο σημείο το οποίο, όπως είπα, είναι το δεύτερο σημείο το οποίο μιλάει για τις ε, για τους φόρους τους δημοσιονομικούς. είναι αν η Βρετανική κυβέρνηση ε, διαπιστώσει μια κατάσταση δεινή σε σχέση με τον προϋπολογισμό και ότι δεν έχουν εκρέψει τα ποσά. Δηλαδή τι θα γίνει. Θα διατεθούν τα ποσά. Γιατί πολιτικά δεν έχω αντίρρηση, ειδικά αν πρόκειται για μια ανθρωπιστική καταστροφή. Θα πρόκειται όμως χρήματα τα οποία διαφορετικά θα πρέπει να ε, επανέλθουν στα κράτη-μέλη ή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Και επίση το σημείο 2, δεύτερο ημισή του, αναφέρεται ότι σε περίπτωση όπου δεν εξευρεθούν αυτά τα ποσά, προτείνουν οι εισηγητές μας, να αντληθούν από τον επερχόμενο προϋπολογισμό του επομένου έτους. Συμβαστική προφορική τροπολογία υπαριθμών 7 πρόταση κανονισμού για το άρθρο 23. Ο εισηγητής λοιπόν προτείνει τα ποσά αυτά να αντιληφθούν όπως είπα από τον προπολογισμό του επόμενου τους. Πολιτικά δεν έχω αντίρρηση, αλλά νομικά δεν μπορώ να είμαι βέβαιος και δεν μπορούμε να είμαστε όλοι, κανείς μας βέβαιος, ε, εάν είναι σύμφωνο αυτό με, τον συνθήκε, με, τον... με τις συνθήκες, με το δίκαιό μας. Αυτό πρέπει να επαληθεύσουμε. για να μην ε, καταρρεύσει όλο το σύστημα. Και επίση το ζήτημα των εμβασμάτων, των λεπτομερών ζητημάτων με, των σχετικών με τα εμβάσματα, τι μεταφορέ, θα ήθελα να εμβαθύνω στα ερωτήματα του κύριου Φέρμ. Οι συνάδελφοι Ριβελίνη και Γκρέσλε στο 1α διατυπώνουν ε, ένα ξεκάθαρο κανόνα και γι' αυτό εδραιώνοντας τον κανόνα αυτό διαγράφουν το β. Το ένα β. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μας διευκολύνει πολύ. Στο ένα δέλτα η δυσκολία που εντοπίζω είναι ότι η διατύπωση που έχει εξευρεθεί ως συμβαστική πρόταση και πρέπει να σας το διαβάσω στα αγγλικά μεταξύ των τμήματων και σημείων που αξιοποιούνται στους σκοπούς για τους οποίους έχουν προσδιοριστεί. Τι σημαίνει σκοπός εν προκειμένου. Είναι σκοπός που απορρέει από την αντίστοιχη γραμμή στον προϋπολογισμό, από την αντίστοιχη θέση στον προϋπολογισμό. Γιατί βέβαια ο καθένας που εκτελεί ένα σχέδιο μπορεί να έχει προθέσεις ή σκοπούς. Και επίσης θα ήθελα εκεί στο DA να ζητήσω μια διευκρίνηση για το τι σημαίνει new quality, νέο χαρακτηριστικό. Τι καλύπτει αυτή η έννοια. Neue Qualität. Άλλο συνάδελφο. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να θέσουν ερωτήματα ή να κάνουν κάποια σχόλια, κύριε Ζεβεράνσκι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για τα χρηματοδοτικά μέσα Άκουσα την παρουσίαση του κ. Ριβελίνη και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Γκάιερ. Η κατάσταση έχει Ο στόχος μας είναι να έχουμε πρόσθετα κονδύλια μέσω των project bonds. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και ας πούμε ότι θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την εξουσία να χρησιμοποιήσει αυτά τα project bonds. Συγχρόνως όμως δεν έχουμε καμία εξουσία ελεγκτική πάνω στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εάν ευσταθεί αυτό λοιπόν, τι θα σημάνει η χρήση αυτών των εργαλείων. Ίσως θα έπρεπε να διοργανώσουμε κάποιο διαγωνισμό για να βρούμε κάποια άλλη τράπεζα η οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτά τα project bonds. Και επίσης το ερώτημα είναι πώς αυτά τα μέσα, τα χρηματοδοτικά μέσα, συνδέονται με αυτά τα οποία έχουν προτείνει οι σοσιαλιστές, δηλαδή τα ευρωομόλογα, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τα σχέδια τα οποία προβλέπονται στα πλαίσια των επερχομένων δημοσιονομικών προοπτικών. Σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές, μετά από αυτά που είπε η κυρία Γκρέσλε, καταλαβαίνω ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της και όλα αυτά. Από τη στιγμή όμως που θα έχουμε μία πρόταση μεταφοράς κονδυλίων μέσα σε μία υποκατηγορία και μετά μέσα σε τμήματα του προϋπολογισμού Μήπως αυτό δίνει υπερβολική ευελιξία στην Κομισιόν. Μέχρι πέρσι θα έπρεπε η Κομισιόν να αντιμετωπίσει το κενό μεταξύ των πιστώσεων υποχρέωσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Και υπήρχε κάθε φορά ένα όλο και μεγαλύτερο επίπεδο μη απορροφουμένων κονδυλίων. Μήπω η δημιουργία μια μεγαλύτερη ευελιξία για την Κομισιόν θα σήμαινε ότι αυτά τα μη δαπανόμενα ποσά θα τύχαναν καλύτερη χρησιμοποίηση ή μήπω θα διατηρούσε την κατάσταση όπω είχε και θα απλώ μείωνε την ελεκτική ικανότητα του Κοινοβουλίου. Το ερώτημα είναι αν το Κοινοβούλιο θα διατηρούσε την ίδια ικανότητα να ελέγχει τα τεκτενόμενα στο δημοσιονομικό χώρο σα. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Ο Γιάνν Μιλντερ αλλά μήπω θέλει κάποιο άλλος να λάβει το λόγο στη συνέχεια. Όχι, μόνο ο Γιάνν λοιπόν. Το είπα προηγουμένω. Εγώ χαίρομαι για την επιμονή της Ingeborg Γκρέσλε. Αλλά έχω και ένα ερώτημα ένα από τα κύρια θέματα συζήτηση για τι επόμενες δημοσιονομικέ προοπτικέ θα είναι το τι θα πρέπει να κάνουμε με τα κονδύλια τα οποία δεν απορροφώνται και δεν δαπανώνται. Εγώ έχω προτείνει μία τροπολογία η οποία θα πρέπει να αποτελέσει και αντικείμενο των συζητήσεων του προπολογισμού για τον επόμενο χρόνο. Η συγγήτρια θεωρεί ότι αυτά θα πρέπει να θεωρούνται ως εισόδημα το οποίο έχει κάποιο προσδιορισμό. Εγώ προτιμώ να έχουμε μια γενικότερη συζήτηση και να πω ότι έχουμε δεσμεύσει κάποια ποσό και υπάρχει ένα ποσό το οποίο μένει ε, θα πρέπει να δαπανηθεί και πάλι για τον ίδιο στόχο. Ίσως όμως αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε σωστή σωστό προσδιορισμό το κονδυλίων, προτιμώ να μπουν σε ένα γενικό αποθεματικό παρά να ξαναγυρίσουν στον ίδιο σκοπό, στην ίδια υποκατηγορία. Άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάποια σχόλια, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Ναι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω εδώ, Νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί στις προηγούμενες παρεμβάσεις καταδεικνύουν κάποιες ανησυχίες τις οποίες συμμερίζεται εν μέρη και η Κομισιόν. Να σταθώ σε δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το θέμα του χρονισμού. Εγώ έχω καταγράψει την κατάσταση ως έχει σήμερα, έχω καταγράψει και το γεγονός ότι η πρόθεση του Κοινοβουλίου ήταν να υπάρξει ψηφοφορία το Σεπτέμβριο για τις τροπολογίες αυτές και για το σχέδιο ψηφίσματος. Για μας αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί έχουμε τονίσει κάθε επανάληψη και κατά συρροή ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε μια πολιτικού χαρακτήρα συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος του 2011. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο διότι εμείς χρειαζόμαστε να έχουμε σαφήνεια για αυτά τα οποία θα ακολουθήσουμε. Θέλουμε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να υπάρχει μια σαφήνεια για το σύνολο των επιμέρους τομεακών προτάσεων ώστε να μπορεί η Κομισιό να παρουσιάσει αυτές τις προτάσεις μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του τέλους του ενεστώτος έτους. Είναι απαραίτητο αυτό για να εξασφαλίσουμε μια συνεκτικότητα μεταξύ της νομοθεσίας κατά τομής και του δημοσιονομικού κανονισμού, το να ξέρουμε ακριβώς λοιπόν σε ποια βάση εργαζόμαστε. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο και ιδίω για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το στόχο της απλοποίησης που έχουμε θεσπίσει όλοι στον εαυτό μας με τον στόχο οι τελικοί αποδέκτες να μπορούν να εργάζονται επί τη βάση κανόνων οι οποίοι θα είναι διαχειρίσιμοι και κοινοί. Το θέμα αυτό λοιπόν του χρονισμού κύριε Πρόεδρε, <clears throat> σας το επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό για την Κομισιόν σε ό,τι αφορά την επίτευξη της αποτελεσματικότητας και όχι για λόγους καθαρής γραφειοκρατίας ή απλώς επειδή θέλουμε να ξεμπερδέψουμε το ταχύτερο δυνατό με ένα θέμα. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Δεύτερη παρατήρηση. Υπήρξαν παρεμβάσεις σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα και σε σχέση με το θέμα των μεταφορών πιστώσεων και κάποιες παρατηρήσεις για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Χρηματοδοτικά μέσα πρώτα. Οι στόχοι που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας, νομίζω όλοι, είναι να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από, τις, ε, από τα κονδύλια που έχουμε στον προπολογισμό με την καταφυγή σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Και όπως είπαν και πολλοί από αυτούς οι οποίοι έλαβαν τον λόγο, είναι σημαντικό τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα να έχουν ένα χαρακτήρα χρησιμοποιήσιμο, διαχειρίσιμο. Αν βρεθούμε με ένα χρηματοοικονομικό ζουρλομανδία σε ό,τι αφορά την διαχείριση αυτών των εργαλείων, θα είναι πολύ περιορισμένη η χρήση των χρηματοδοτικών αυτών μέσων. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα λοιπόν, αυτό γίνεται διότι σε ορισμένε περιπτώσει, και σκέφτομαι εδώ πέρα του, τα ευρωομόλογα τα οποία αναφέρθηκαν, ή τα project bonds καλύτερα, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να θεραπεύσουμε <clears throat> τις ελλείψεις που παρουσιάζονται σε επίπεδο αγορών. Εμείς εργαζόμαστε με αγορές με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. που η κύρια μέρημνά τους είναι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια. Αυτό λοιπόν που η δημόσια χείρ μπορεί να προσθέσει εδώ είναι μια ενίσχυση της ασφάλειας ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το χάσμα που επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα υποδομών να υπάρχει μια παρέμβαση του δημοσίου τομέα και σκέφτομαι τα project bonds χάρη στις εγγύσεις που μπορεί να δώσει ο κοινοτικό προπολογισμό και πάντα μέσα στα όρια τα οποία προβλέπει ο κοινοτικό προπολογισμό, είτε μέσα από πιο κλασικά χρηματοδοτικά μέσα όπως αυτά που αναφέρθηκαν στη συζήτηση αυτή. Και θα ήθελα σχετικά να σας πω ότι υπήρξε <clears throat> και μνήμα ορισμένων μέσων τα οποία δεν έχουν φαίνεται λειτουργήσει πολύ καλά Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαμεμοιρασμένης διαχείρισης που είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ότι στην περίπτωση της άμεσης διαχείρισης γιατί στην περίπτωση αυτή, ιδίω τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ανάγκη για πολλά κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες για να μπορούν πράγματι να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα προσχώματα λοιπόν αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί έχουν σε μεγάλο βαθμό αρθεί. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες των τροπολογιών που έχουν να κάνουν με τα χρηματοδοτικά εργαλεία ή μέσα. Το μήνυμα που θέλω να δώσω όμως σε αυτό το σημείο είναι κάτι το οποίο συνάδει πολύ με αυτά που είπανε πολλοί παρεμβαίνοντας. Δεν πρέπει να έχουμε ακαμψίες. Σεβόμεθα απόλυτα το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει τη δυνατότητα του ελέγχου και της εξέτασης της χρησιμοποίησης των κονδυλίων που ετέθηκαν σε εφαρμογή. Αν όμως η προσέγγιση η οποία θα επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οδηγεί στην ακαμψία, τότε ας τα ξεχάσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν θέλουμε να έχουμε εργαλεία τα οποία από τη μία πλευρά εμπεριέχουν κίνδυνους και από την άλλη μεριά ακαμπτοποιούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν λειτουργούν έτσι οι αγορέ. Και υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, κάποιες πρόοδοι οι οποίες <clears throat> επετέθησαν στον τομέα των μεταφορών πιστώσεων. Αλλά εγώ θέλω να επανέλθω σε ένα ερώτημα το οποίο είχαμε συζητήσει κάτι επανάληψη στο παρελθόν. Γιατί μέσα στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να επανέλθουμε σε διατάξεις οι οποίες είχαν εξαφανιστεί. Ε, και τις είχαμε απλουστεύσει, οι οποίες είχαν ήδη εφαρμοστεί με οριζόντιο τρόπο, οι οποίες ήταν ικανοποιητικές για όλους. Εμείς από πλευράς Κομισιόν πραγματικά δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να επανέλθουμε στις ε, έξι εβδομάδες όταν έχουμε τρεις εβδομάδες. Και με τις τρεις εβδομάδες όλοι ήταν ικανοποιημένοι. Ενώ η ιστορία των ε, μεταφορών πιστώσεων μας δείχνει ότι αν κοιτάξουμε τα δέκα τελευταία χρόνια ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα. Για δεκάδες επί δεκάδων μεταφορών πιστώσεων υπήρχε μόνο δυσκολία σε τρεις α, μεταφορές, δηλαδή ανθιπολεπτομέρειες σε σχέση με τον τεράστιο όγκο των, του αριθμού, τον τεράστιο αριθμό των πιστώσεων των μεταφορών πιστώσεων που έγιναν. Εάν επανέλθουμε σε έξι εβδομάδες Πού είναι η απλούστευση. Τώρα, για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Υπάρχει πρόοδος, πρέπει να σεβαστούμε τους όρους της ε, κοινή ε, συνεννόησης που, και συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω, Πρόεδρε, για το θέμα αυτό. Από πλευράς Κομισιόν, επαναλαμβάνω, μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε όσο μπορούμε στις εργασίες σας και χαίρομαι που βλέπω ότι γίνεται πραγματική συζήτηση για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα σας βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε και εσάς αλλά και το Συμβούλιο, ούτω ώστε να πλησιάσουν οι μεν τους δε, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο με βάση το ρόλο που έχει η Κομισιόν στα πλαίσια της διαδικασίας της συναπόφασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζουανζόν. Βλέπω τη γλώσσα του, του σώματος ορισμένων συναδέλφων και βλέπω ότι ορισμένοι ενοχλήθηκαν. Μερικές φορές το πρόσωπο της κυρίας Γκρέσλερ συσπώνταν με έναν τρόπο που ήταν πολύ εύγλωτος. Λοιπόν, για να αποφύγουμε το χάος, τέθηκαν πολλά ερωτήματα. Θέλουμε ε, απαντήσεις σε 8 σημεία. Ε, κύριοι συνεισηγητές, πολλές ερωτήσεις για τα, τη σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου δικαίου, για τα θέματα μεταφοράς πιστώσεων, για τα θέματα της κατεξουσιοδότηση πράξεων, για τα θέματα της διαφάνειας για τη σύγκρουση συμφερόντων. Ο κύριος Μούλτερ μας ζήτησε τι πρέπει να κάνουμε με τα μη ε, δαπανημένα κονδύλια. Επίσης, η κυρία Μπραντνερ έκανε μια ερώτηση για τον κατάλογο ψηφοφορίας και τι θα γίνει με το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας. Τι θα γίνει, ας πούμε, την ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Ο κύριος Φέρμ ρώτησε επίσης τους εισηγητές αν θέλουν συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ναι ή όχι. Νομίζω ότι συνόψισα όλες τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Η... Ποιος ε, εισηγητής θέλει πρώτος να παρέμβει, η κυρία Γκρέσλερ. Ο κυρίας πρώτες. Μάλιστα. Α μιλήσουμε λοιπόν για τι παλιέ ιστορίε. Να να συζητήσουμε τον κύριο Φέρμ το θέμα τη διαδικασία. Καταρχά, εμεί ω ηγητέ, πολύ ευχαρίστω να συζητήσουμε κάθε θέμα. Όντω πιέζει ο χρόνο, αλλά ο κύριο Γενικό Διευθυντή πιστεύω δεν μπορεί να αποκρύψει την κατάσταση, τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή χρονιά. Δεν μπορεί δηλαδή να κλείσουμε όπως πρέπει την χρονιά εγκαίρως. Άρα το θέμα δεν είναι ο χρόνος τόσο. Εμείς δεχόμαστε κάθε πρόταση να συζητήσουμε. Είναι ζήτημα, όπως έχουμε πει, και ε, σωστής και ακριβοδίκαιης μεταχείρισης να δεχόμαστε τις προτάσεις των συναδέλφων. Εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ ως λύση μια ε, δεύτερη ανάγνωση για να δούμε ε, τι σκέφτονται οι συνάδελφοι και να μεταφέρουμε στο Συμβούλιο τις θέσεις αυτές. Γιατί θα δείτε ότι και στο συμβαστικό πακέτο υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, που έχει είτε καταγράψει ο κύριος Μπέγκε στο, από το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, είτε ο κύριος Μίλντερ είτε η Γραμματεία έχουν προτείνει. Είναι δύο δηλαδή διαφορετικές τροπολογίες μεταξύ ε, των συναδέλφων αυτές που κατετέθησαν και τις οποίες δεχτήκαμε. Είτε λοιπόν ε, πούμε ότι πρόκειται για ποσά τα οποία είναι γενικές δαπάνες ή ειδικέ δαπάνες, σε πάση περιπτώσει έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να συμπεριλάβουμε, για να δεχθούμε στο κείμενο της απόψης των συναδέλφων. Και δεν μας ε, φοβίζει η μάχη που έχουμε μπροστά μας, όσο δύσκολη και αν είναι. Άλλωστε δεν πρόκειται για μάχη που διεξάγεται έναντι των συναδέλφων. Έχουμε απλώς έναν αγώνα στον οποίο να αποδιόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και με ανοιχτό πνεύμα. Διπραγματευόμαστε λοιπόν με το Συμβούλιο, κοιτάμε τι μπορεί να γίνει δεκτό, τι δεν μπορεί να γίνει δεκτό και στο βαθμό του δυνατού προχωρούμε σε ταχύ ρυθμού, εφόσον είναι δυνατό αυτό. Αν και όπως είπα για το πολιτέ, δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι πάντα δυνατό, ε, λόγω ακριβώς της δυσκολία του θέματος. Και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται πάνε όλο και πιο περίπλοκα να γίνουν, ε, όχι να απλουστευτούν. Άρα κύριε Φέρμε, πολύ ευχαριστώ να συζητήσουμε τις προτάσεις σας. Για τα δημοσιονομικά μέσα τώρα. Να συνεχίσω. Έχουμε δημοσιονομικά μέσα αποθηκευμένα σε φορολογικούς παραδείσους. Και γι' αυτό ζητώ να γίνει κάποια εποπτεία γιατί όπως θα δεν γνωρίσουμε τώρα τίποτα για τα όσα συμβαίνουν, η Επιτροπή η ίδια μπορεί να δώσει τις ε, πληροφορίες. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπους μπορεί να αντλήσει πληροφορίες, μόνο και μόνο επιταδεύουν ότι εκατομμύρια προέβλεπαν κάποιο τύπου εποπτεία των δημοσιονομικών μέσων. Μην ξεχνάμε ότι εδώ πρόκειται για 5 δις ευρώ. Και είχαμε τη χαρά ε, στο έτος 2010 στην απαλλαγή να δούμε πόσο σημαντικά ποσά και πόσο χαμένα ήταν αυτά τα σημαντικά ποσά. Άρα λοιπόν, ε, και επειδή είδα και ένα non-paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με βάση και τα έγγραφα της Επιτροπής, για τα οποία όμως δεν είμαι καν βέβαιη εάν εντοπίζουν το πρόβλημα στι. σωστές του διαστάσεις. Γιατί διότι φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σερβίρει στο, κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι στο Κοινοβούλιο. Έστω και άτυπα δηλαδή. Εγώ έχω δει κάποια στοιχεία τα οποία δεν έφτασαν ποτέ επισήμως στο Κοινοβούλιο από πλευρά τη Επιτροπής. Για δε τι ε, μεταφορές κονδυλίων. Να το συστήσουμε και διμερώς αν προτιμάτε. Το 7 που λέμε αναφέρεται μόνο στον προϋπολογισμό και όχι, μόνο, και όχι στα υπόλοιπα. Όχι τα ποσά δηλαδή τα οποία πάνε και έρχονται στο τέλος του ε, έτους ε, γιατί κάπου κάτι δεν λειτουργήσε σωστά. Το 7, η τροπολογία 7, έχει να κάνει με τον παλαιό δημοσιονομικό ε, κανονισμό τον οποίο χρησιμοποιούμε σε, αυτό το, σε αυτή τη διατύπωσή του για να ρυθμίσουμε καινούρια στοιχεία. Προσπαθούμε από τα δεδομένα που έχουμε τώρα, από τις δυνατότητες που έχουμε τώρα, να προχωρήσουμε προς μία απλούστευση, που είναι ο στόχος τον οποίο τίνουμε, το στόχος τον οποίο επιδιώκουμε. Και εδώ αλλάζει, ε, πέραν των ποσοστών κτλ., η ιστορία των έξι εβδομάδων. Εμένα μου φαίνεται ότι τρεις εβδομάδες δεν αρκούν για να βουλευτεί να δει ε, τέτοιου είδους ε, λογαριασμού. Αν υπολογίσουμε εδώ και τις οπωσδήποτε δεν αρκούν. Γι' αυτό ζητούμε την επέκταση, την παράταση αυτή τη προθεσμίας στι έξι εβδομάδε. Και λέμε επίση ότι η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζει η Επιτροπή είναι η μετάφραση για να έχουμε τα έγγραφα εργασία ή σε όλε τι επίσημε γλώσσε, τουλάχιστον στι τρει γλώσσε εργασία. Πάντω αυτό θέλουμε να απλουστευθεί. Τα έγγραφα info της Επιτροπής. Είναι τα ενημερωτικά έγγραφα για τις μεταφορές κονδυλίες. Τώρα, για να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των άρθρων 23 και 24 που ζητάτε. Εμείς εγκαταλείψαμε το άρθρο 24 γιατί εκεί γινόταν η αναφορά στην ε, συμφωνία του 2009 ε, και τα 100 εκατομμύρια των πληρωμών. Γι' αυτό λέμε ότι θα μπορούσε καταρχάς να αποσταλεί ο λογαριασμός και εκ των υστέρων να εγερθεί η ένσταση ή η ε, μομφή για να προχωρήσουμε κάπως πιο γρήγορα. Να έχω την ευκαιρία δηλαδή να αμφισβητήσω μία πρόταση εφόσον κάτι δεν μου αρέσει. Αλλιώ το έγγραφο, το, το έγγραφο του Κοινοβουλίου για την μεταφορά των κονδυλίων έχει κατευθεί από 21η Ιουνίου. Όπω βλέπετε, εμεί πάντα έχουμε κάνει γέρο στη δουλειά μα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω για όλου του συναδέλφου τη σημασία αυτού του εγγράφου που κρατάω, διότι είναι πολύ ε, σημαντική η διαφορά μεταξύ των όσων ίσχυαν μέχρι το 2009 και των στοιχείων που έχουμε έκτοτε ε, να χειριστούμε και των στόχων που επιδιώκουμε, δεδομένου ότι έχουμε και εντατικοποίηση της εργασίας μας. Η πρόταση λοιπόν για το 2010 εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε, στον τίτλο, σε, στο τμήμα που αφορά μια συγκεκριμένη γενική διεύθυνση, μπορεί να ε, μεταφέρει κονδύλια εφόσον υπάρχουν. Μέσα όμως στο, στο τμήμα αυτό που αφορά τη συγκεκριμένη γενική διεύθυνση. Αυτό αποτελεί μια σημαντική διεύρυνση αρμοδιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εν τη αυτή περίπτωση πιστεύω ότι εάν δεν κάνουμε λίγη παραπάνω προσπάθεια στον προπολογισμό για να ρυθμίσουμε τα πράγματα όπως πρέπει, ας μην κάνουμε και τίποτα στη τελευταία ανάλυση, ας μην συντάσσουμε προϋπολογισμούς. Γιατί βγαίνουμε στην Ολομέλεια, ε, αντιπαρατηθέμεθα με το Συμβούλιο και μετά μας λέτε εκ των υστέρων δεν μπορούμε να κάνουμε καμία επαλήθευση. Ε, δεν γίνεται αυτό, δεν έχει καμία ε, αξία όλη μας η προσπάθεια και γι' αυτό καταλήγω εγώ στο λογικό συμπέρασμα ότι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε ουσιαστικά τον έλεγχο. Το Common Understanding, το Μνημόνιο Συνεννόηση, ήταν μια συμφωνία μεταξύ των νομικών υπηρεσιών, δεν πέρασε ποτέ από την Ολομέλεια. Πέρασε από την Ολομέλεια μόνο η έκθεση Σάιερ, την οποία ψηφίσαμε με πλειοψηφία 95% συντριπτική πλειοψηφία και που ξεπερνά σε μεγάλο βαθμό το πεδίο τη ε, Common Understanding του, του Μνημονίου Συνεννόηση. Και παρακαλώ του συναδέλφου να το ξαναδιαβάσουν το Μνημόνιο αυτό Συνεννόηση, συνάδελφοι, προσεκτικά, διότι δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα, δεν αγγίζει καν τα προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μα. Στο σημείο 2, επί παραδείγματι, αναφέρει κάποιε επιλογέ ε, ω προ το ζήτημα για το πόσο θα πρέπει να διαρκέσει αυτή η πράξη ε, εξουσιοδότησης. Εμείς λέμε ότι η εξουσιοδότηση θα πρέπει να διαρκεί τρία χρόνια. Το έχουμε ήδη αποφασίσει αυτό. Ε, και λέμε ότι και αποφασίσαμε εκ των υστέρων ότι θέλουμε για να υπάρχει μια ομοιόμορφη ρύθμιση όλων αυτών των πράξεων συνεννόηση, να υπάρχει αναθεώρηση τα τρία χρόνια και η επαλήθευση κτλ. Δεν θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια απεριόριστη εκχώρηση των εξουσιών αυτών. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα γίνει και στι δύο περιπτώσει ε, ω προθεσμία, ω όριο μάλλον ε, ισχύω ή τριετία. Για να υπάρχει μια συνέπεια στο μνημόνιο συνεννόηση και, το συζήτησαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Λένε, τον πρόεδρο τη Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, διεξοδικά για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθο. Δεν επιλύει κανένα πρόβλημα. Προσπαθώ αυτό το πίνακα εδώ να τον καταρτήσω λέγοντα τι μα λέει το μνημόνιο συνεννόησης, τι μα λέει η πρόταση επιτροπή, τι μα λέει η δική μας η πρόταση στο κάθε σημείο, μαζί με μια, ε, με μια υπόμνηση για την διαδικασία της συναπόφασης που έχει επισημάνει η νομική μας υπηρεσία, δηλαδή έτσι ώστε να μην ξεπερνούμε τα απολύτως αναγκαία ως αρμοδιότητες στη δραστηριότητά μας Και δεν θέλω το μνημόνιο συνεννόησης να χρησιμοποιείται ως ένα επιχείρημα ότι, το οποίο τελικά θα οδηγεί σε νέκρωση όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να φέρει καρπούς, όχι να είναι τελικά αρνητική η επίδρασή του. Φραντσέσκα, για την παρατήρησή σου θα σου απαντήσω με το email για τις ε, προτάσεις ε, για, τις, ε, για την τροπολογία που έλεγες. Είχα μια συζήτηση επί μακρόν για τα θέματα της γεωργίας και τα γεωργικά ταμεία και το κατά πόσον θα έπρεπε να κοινοποιούνται τα στοιχεία αυτά ή όχι. Και θα ήθελα να σου πω ότι υπάρχει μια απόφαση για το θέμα της δημοσίευσης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βάσει οποίας οφείλουμε να προχωρήσουμε, και έχουν βέβαια και τη σχετική ευθύνη οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να περιμένουμε μέσα σε κάθε περίπτωση να μην χάνεται από το ένα στάδιο στο άλλο κάτι που έχει κερδιθεί στο παρελθόν. Ο συνάδελφος Λιμπεράτσικη και επίσης ε, διατύπωσε πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις και τον ευχαριστώ ως συνήθως κάποια ζητήματα μας αναγνωρίζουν, κάποια, οι τομείς μας αναγνωρίζουν μόνο πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες κύριε Ριμπεράτης και θα πρέπει να σας πω και θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς ε, εάν θέλουμε να παραχωρήσουμε, να εκχωρήσουμε και άλλους ε, τομείς αρμοδιοτήτων ή εξουσιών. Εν πάση περιπτώσει, αν, αν μπορούσαμε μέχρι τις διακοπές να συμφωνήσουμε για τις συμβαστικές τροπολογίες, μπορούμε και μέσω του email να συνεργαστούμε. Εγώ πάντα, ακόμα και στις διακοπές, μου παρακολουθώ το ηλεκτρονικό μου ταχυδραμείο και έτσι αν συντονίσουμε τις προσπάθειές μας το Σεπτέμβριο και στην πρώτη ολομέλεια ακόμα του Στρασβούργου μπορούμε να ε, προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριβελίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κυρία Γκρέσλερ ήταν πολύ σαφής στις απαντήσεις που έδωσε. Και μίλησε και για κάτι σοβαρό. Αναβάλαμε για, την, για το Σεπτέμβριο την ψηφοφορία. Έχουμε όλο το χρόνο για να εμβαθύνουμε κάποια θέματα λοιπόν. Και μέσω email. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις για τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την τελευταία διαπίστωση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όπου για τα δημοσιονομικά εργαλεία μας είπε να μην ε, βάλουμε τσουρκλωμανδία, όπως είπε η Επιτροπή, στα χρηματοδοτικά μας, τα οποία θα πρέπει να είναι απλά, ε, χρήσιμα και να λειτουργούν τάχιστα. τάχιστα. Εγώ διερωτώ με, δεν υπάρχει μια τρίτη οδός ανάμεσα σε μια ε, γρήγορη διαδικασία και σε, που μπορεί να έχει τον κίνδυνο της πλήρους αναρχίας. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλερ και ζητάω από την Κομισιόν να επικαιροποιήσει αυτό το παλιό ε, non-paper του 2010, ούτω ώστε να στείλει στο Κοινοβούλιο ένα πλαίσιο πιο ξεκάθαρο για το πώς θα επενδυθούν τα χρήματα ε, με τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να σας βάλουμε ζουρλομανδία, αλλά δώστε μας σωστά στοιχεία για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Γιατί αλλιώς δεν μας δίνεται τη δυνατότητα να εργαστούμε σωστά. Περιμένω λοιπόν και εγώ και η κυρία Γκρέσλερ το συντομότερο δυνατόν αυτή την επικαιροποίηση του non-paper. Τώρα, για τα κονδύλια, για τις πιστώσεις. Μην ξεχνα... Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους λόγους για τους οποίους είπαμε το η τάδε πίστοση για τον τάδε σκοπό. Δεν είναι δεδομένο ότι ο σκοπός αυτός ήταν λαθασμένος και ότι είναι ξεπερασμένο και ότι δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι είναι χρήσιμο να επιβεβαιώσουμε αυτόν τον προσδιορισμό για να μην τιμωρήσουμε αν θέλετε κάποιες ε, περιφέρειες, κάποιες περιοχές ε, που μπορεί να στερηθούν ε, κονδύλια έτσι αν αλλάξουμε προσδιορισμό. Επίσης, συμφωνώ με τον συνάδελφο που είπε ότι ο συμβασμό 7 άρθρο 23 θα πρέπει να το, αυτό το σημείο να το ψάξουμε περισσότερο για να δούμε κατά πόσο συνάδει με τη συνθήκη. Για την ψηφοφορία επίσης. Συμφωνώ με τη συνάδελφο. Ίσως πρέπει να, πλήσου, να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε πρώτη ανάγνωση και να ψηφίσουμε πλήρως για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλύτερα εν συνεχεία. Για τα υπόλοιπα θέματα νομίζω ότι η κυρία Γκρέσλερ απάντησε με αρκετά ακριβή τρόπο. Τώρα για τις μεταφορές πιστώσεων. Στην πρότασή μας υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ μιας ε, επιτάχυνσης εφαρμογής της διαδικασίας και μεταφορών πιστώσεων που έχουν πιο πολιτικό χαρακτήρα. Έχουμε κάνει μια διαφοροποίηση. Φυσικά μπορούμε να ακούσουμε εδώ διάφορες ιδέες από τους συναδέλφους, διάφορες συμβουλές αν θέλουν να μας δώσουν για αυτή τη διαφοροποίηση των πιστώσεων. Ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί πήραν απάντηση στα ερωτήματά τους. Είσαστε όλοι ικανοποιημένοι. Μια τελευταία παρατήρηση κυρία Γκρέσλε. Το ελεγκτικό συνέδριο θα ήθελε πράγματι να ρωτήσει τι έχει γίνει ακριβώς με το, την εφαρμογή του 2010. Εγώ δεν έχω δει εδώ πέρα καθόλου στοιχεία σχετικά. Κοιτάζω προς το ελεκτικό συνέδριο. Είχαμε ρωτήσει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλατε να απαντήσετε το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι κατάλαβα αναφέρεστε στον κανονισμό του 2010. Μήπως μπορεί κυρία Γκρέση να επαναλάβει το ερώτημα, παρακαλώ. Κυρία Γκρέση, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε. Οι εμπειρίες μας με το χρηματοδοτικό εργαλείο το 2010 είναι να δούμε τι ακριβώς προέκυψε. Εμεί θέλουμε να ξέρουμε αν είναι σωστή η νομοθεσία μα. Καταλάβατε, έχετε παρακολουθήσει το ηλεκτρικό συνέδριο. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι μια γενική παρατήρηση. Πολλές από τις τροπολογίες εδώ έχουν να κάνουν πολιτικές εξαρτήσεις για τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για το ελεκτικό συνέδριο είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο λογοδοσίες για τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία. Επομένως, το γεγονός ότι πρόκειται να υπάρξει κάτι στο δημοσιονομικό κανονισμό το οποίο να διέπει την χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων και την λογοδοσία για αυτά είναι κάτι το θετικό. Όπως είπε όμως και το ελεκτικό συνέδριο στη γνωμοδότησή του, αυτό δεν είναι ένα τεράστιο βήμα. Θα θέλαμε να έχουμε ένα πιο σαφές πλαίσιο, ώστε, όπως είπε και η κυρία Κλέστε, να είναι σαφές για ποιο χρονικό διάστημα τα χρήματα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια στιγμή περνάνε στα χέρια του τελικού αποδέκτη. Επομένως, σε ποιο σημείο θεωρούνται αυτά τα κονδύλια ότι έχουν δαπανηθεί. Εδώ υπάρχει φυσικά μία διαφορά γιατί τα χρηματοδοτικά εργαλεία δημιουργούν στοιχεία ενεργητικού και δεν απλώς εκταμίευση χρημάτων. Οπότε το, το δημοσιονομικό πλαίσιο εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο. Και επίσης θα θέλαμε να ξέρουμε και περισσότερα για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη χρήση αυτών των ε, δημοσιονομικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Τι γίνεται με, την, με το λεγόμενο common understanding. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα θέλαμε να έχουμε η εμπειρία μας είναι ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Επομένως όλες αυτές τις προτάσεις για το νέο δημοσιονομικό κανονισμό είναι απόλυτα καλόδεκτες από εμάς. Θα θέλαμε να εξερευνηθούν περισσότερο. Βλέπω η κυρία Γκρέσεν να ανέβει. Καταφατικά δεν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην ζήτηση αυτή. 29 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Ριβελίνη. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Τις τελευταίες μέρες κάθε φορά λέγεται κάτι διαφορετικό. 22, 23, 26 Σεπτεμβρίου, 29. Πέστε μας ποια είναι η στιγμή που θα γίνει συζήτηση για να μπορούμε να είμαστε ενήμεροι. Το πρόβλημα, λέει ο κύριος Στάση, είναι ότι η γραμματεία μας προσπαθούσε να βρει μια ημερομηνία η οποία θα βόλευε και τους δύο εισηγητές. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε διότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι παρόντες οι δύο συνεισηγητές στη στιγμή της συζήτησης. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρότεινα εγώ είναι να βρούμε πρώτα μια κατάλληλη ημερομηνία και μετά θα σας ενημερώσουμε με email και τότε μπορώ να σας πω ότι θα είναι αυτή η οριστική ημερομηνία. Κλείνει λοιπόν η κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών προπολογισμού και ελέγχου του προπολογισμού. Θα περάσουμε τώρα και πάλι στην ημέρηση διάταξη της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. αφού όμως κάνουμε μια σύντομη διακοπή, ώστε αυτοί που θέλουν να φύγουν να μπορέσουν να αποχωρήσουν.